Everyone, if you want to take your seats, then maybe... Καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει 10 λεπτά σε σχέση με την προβλεπόμενη για σήμερα το μεσημέρι ώρα έναρξης. Θα σας ε, πω τα όσα λέω συνήθως ε, πιο μετά. Θα ξεκινήσουμε το σημείο της ημερησιάς διάταξης ε, που είναι ακρόαση του υποψηφίου για θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΚΑ. που είναι στο επίκεντρο της σημερινής μας ημερήσιας διάταξης, εφόσον το πρωί είχαμε την ακρόαση και τώρα συνεχίζουμε Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι ο τελικός διευθυντής ε, θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση κατάλογο ψηφιότητων που πρότεινε η Κομισιόν μετά από πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιστοσελίδες και σε άλλες εφημερίες περιοδικά. Πρέπει να έχει εμπειρία, να έχει διοικητικές δεξιότητες, ιδίως εμπειρία στα χημικά, ε, την ασφάλεια και τα σχετικούς κανονισμούς. Πριν όμως ε, οριστεί, πρέπει να προσέλθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Για να έχουμε μία ακρόαση με τον ε, υποψήφιο τον κύριο Μπιέρν Γιάν Χάνσεν. Θα τον ακούσουμε και θα συζητήσουμε μαζί του. Είναι ο υποψήφος που επελέγει 28-29 Σεπτεμβρίου. Κύριος Χάνσεν ε, ήταν επικεφαλής μονάδας ε, ασχολείται με βιώσιμα χημικά προϊόντα από την ε, Διεύθυνση Β της Γενικής Διεύθυνσης Σχετικής του Κομισιόν από το 2012 είχε αυτή τη θέση και θα έχει πενταετή θητή εφόσον εκλεγεί στη νέα του θέση. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Χάνσεν για να μας πει τα δικά του για 10 λεπτά και έπειτα θα έχουμε μία ανταλλαγή ρωτήσεων απαντήσεων. Θα διαρκέσει 25 λεπτά και οι υπόλοιποι 3 λεπτά. Μάλλον η πρώτος γύρος ο κάθε ομιλητής για την απάντηση και την ερώτηση θα έχει 5 λεπτά στη θέση του και στο δεύτερο γύρο 3 λεπτά. Λοιπόν, καταρχάς ο κύριος Χάνσεν να πάρει το λόγο και να μας κάνει την παρουσίασή του. Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα, αλλά ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να σαραστούμε λοιπόν και στη συνέχεια για θέματα που μας ενδιαφέρουν ως Επιτροπεριβάλλοντος. Ε, ευχαριστώ πολύ, εξότιμη κυρία Πρόεδρε, εξότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάθομαι εδώ ε, μπροστά σας για να σας ε, κάνω αυτή τη δήλωση και βέβαια πως βλέπω στη συνέχεια στο γύρο τα απαντήσεων και στην συζήτηση που θα επακολουθήσει και βέβαια και στη μελλοντική συνεργασία που ελπίζω να έχουμε εφόσον οριστώ σε αυτή τη νέα θέση. Εν είδη αγωγής, θα σας πω δύο λόγια για εμένα και να εξηγήσω ποια είναι τα κίνητρα που με παρακίνησαν ε, να υποβάλω ψηφάτη για τη θέση αυτή, την οποία επιθυμώ σφόδρα να αναλάβω και γιατί μπορώ να σας, πώς μπορώ να σας πείσω ότι πραγματικά είμαι κατάλληλος για αυτή τη θέση. Είμαι δανός, υπήκος, αλλά 11 ε, χρόνια μόνο τη ζωή που τα έχω περάσει στην ε, Δανία, τα 11 τα έχω περάσει, μάλλον 13 στην Ιταλία, 13 στο Βέλγιο, 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 στη Γερμανία, 1 χρόνο στη Φιλανδία. Αν προσθέσετε θα βρείτε και την ηλικία μου. Είμαι επιστήμον, σπούδασα στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες, πήρα μάστερς, έχω μπάτσελο στα μαθηματικά, στην ε, ε μαθηματικών μοντέλων και οικονομικά πήρα ε, μετεπένων και έχω και PhD από την Ολλανδία, από το Eindhoven, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο, στα μαθηματικά, θεωρία πιθανότητων. Έπειτα ακολούθησα για κάποιο καιρό μια ακαδημική σταδιοδρομία, αλλά για 26 χρόνια εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των χημικών. Κατά το ίμιση της καριέρας μου στο επιστημονικό κομμάτι και κατά το δεύτερο ήμιση στο πολιτικό κομμάτι. Εξού και θέτω υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, εξού και το πάθος μου να αναλάβω αυτή τη θέση. Θέλω να είμαι μια διαπαφή μεταξύ πολιτικής και επιστήμης. Αυτό με συναρπάζει, πόσο δε μάλλον για τον τομέα των χημικών, που ποτέ δεν βαριέσαι, πάντα έχεις να αντιμετωπίσεις μια νέα πρόκληση, ένα νέο πρόβλημα και όταν το επιλύεις αυτό το πρόβλημα, αυτή την πρόκληση, δεν, είναι, ε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ε, και ήμουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 χρόνια. Αλλά εργάστηκα λίγο πολύ πάνω στα ίδια ζητήματα. Με το ίδιο πάθος λοιπόν ε, θα εργαστώ και στη συνέχεια και θέλω να μιλήσω τώρα για τις δυνατότητες. Οι ικανότητες μου έχω δει το επιστημονικό, τεχνικό, πολιτικό ε, σκέλος και εδώ στις ε, όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι. Επομένω γνωρίζω πολύ καλά πώς ε, θα μπορέσουμε να παντρέψουμε επιστήμη και πολιτική. Και επίσης ε, γνωρίζω πώς μπορώ να τα παντρέψω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω εργαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε επίπεδο ΣΑ και στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, όπου συμμετείχα σε ομάδες εργασίας ε, τεχνικές, ε, συμμετείχα και στη σύμβαση της ε, Οκχόλμης, παρασκευαστικές εργασίες για το επίμους οργανικού ρήπους και εδώ στις Βρυξέλλες ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπείας για να στο κόλμη Βασιλεία της συμβάσης αυτής τρεις φορές με επικεφαλής της αντιπροσωπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι έχω καταφέρει να μάθω να διαχειρίζομαι το περιεχόμενο της εργασίας μου στα διάφορα μου καθήκοντα από desk officer μέχρι αναπληρωτής ε, διευθυντής, ματάρχης, ε, διευθυντής κτλ διαχειρίζομαι όχι μόνο βέβαια το εργατικό δυναμικό, αλλά και το περιεχόμενο της εργασίας. Με αυτές τις ικανότητες ελπίζω να βλέπετε και εσείς, ελπίζω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις που σίγουρα έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα πέντε χρόνια το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει πάντοτε ενδιαφέρουσες προκλήσεις να μας προσφέρει, όπως ε, ισχύει και για την επόμενη πενταετία. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για το 2020-2025 που προσταποδεύει η Ευρώπη. Έχουμε το ζήτημα του Brexit. Επίσης έχουμε και να ε, φροντίσουμε η ΕΚΑ, το προσωπικό της, ε, οι δεξιότητες, οι ικανότητες που έχει συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με το νομοθεσία στον τομέα των χημικών ουσιών να μπορεί να είναι υποφελία της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό θεωρώ ότι δικές μου δεξιότητες, ικανότητες και το υπόβαθρο που έχω ε, μπορεί να είναι χρήσιμα εδώ ε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τους συναντέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω απ' όλα βέβαια για την ΕΚΑ και το προσωπικό της. Αυτό που θέλω πάνω απ' όλα είναι να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το δυναμικό της ΕΚΑ και για να προωθήσει ακόμη περισσότερο την υλοποίηση της νομοθεσίας για τα χημικά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω επειδή έχω υπόψη ότι ο χρόνος είναι λιγοστός και δεν ε, εξάντλησα τον χρόνο που είχα στη διάθεση μου, το δεκάλεπτο δηλαδή, πρόεδρος. Θα ξεκινήσει λοιπόν τώρα ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση, ένα ερώτημα, η δευτερολογία, ε, μάλλον ένα λεπτό δευτερολογία, ερώτηση-απάντηση. Δύο λεπτά δηλαδή συνολικά, πέντε ο κάθε ο πρώτος είναι ο κύριος Νόρμπερτ Λίνς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Μια και έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να περάσω κατευθείαν στην ερώτησή μου. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του κανονισμού για τα βιοκτώνα και το ρόλο που θα έχει η ΕΚΑ σε αυτό. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι οι διαδικασίες για την αδειοδότηση, πώς θα εγκριθεί μια ουσία για να εγκριθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σε δεύτερο επίπεδο ένα βιοκτόμονο που έχει εγκριθεί πώς θα προχωρήσει σε παιδοκρατών μελών χωρίς να επιβληθούν υπερβολικές δαπάνες για τον ε, παραγωγό. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρές, αλλά και τον όταν πρόκειται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα σας ε, παρουσιάσω πρώτα τα γενικά βήματα που προβλέπει ο κανονισμός για τα βιοκτώνα, που είναι αντίστοιχα με αυτά του κανονισμού για τα οκτώνα. Και μετά θα αναφερθώ στην δεύτερη ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο, δύο στάδια στη διαδικασία. Λοιπόν, η έγκριση της ενεργού ουσίας, με τα δεδομένα που δίνουν οι, οι σχετικές εταιρείες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν τα κράτη εισηγητές να αξιολογήσουν και να υποβάλουν τα πορίσματά τους στην υπηρεσία μας, η οποία μετά επαληθεύει τα δεδομένα αυτά, βάσει της οποίας επαλήθευσης μπορεί να καταχωρήσει ως συγκεκριμένη ή μη την ενεργό ουσία. Η αξιολόγηση αυτή σημαίνει ότι υπάρχει μια χρήση μέσα από την οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι η ενεργός ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ασφαλή. Πρέπει δηλαδή η μία χρήση να χαρακτηριστεί ως ασφαλής για να καταχωριστεί στις συγκεκριμένες η ενεργός ουσία. Το δεύτερο στάδιο είναι η έγκριση προϊόντος που εδώ διαφοροποιείται ο κανονισμός των βιοκτωρών από αυτών των ζυζακτιωτώνων, μια διαδικασία έγκρισης του προϊόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αλλά και δυνατότητα αυτό να γίνει από τα κράτη-μέλη. Εάν Υπάρχει ζήτημα μεταξύ κρατών μελών, η όποια διαφορά ως προς τη διαδικασία διοδότησης μπορεί να επιληφθεί με, να έναν, ένα μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης. Αυτή είναι η διαδικασία. Βεβαίως η ερώτησή σας είναι ότι μπορεί μια τέτοια διαδικασία να είναι αρκετά δαπανηρή και να ε, φέρει σε δυσκολία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα καλούνται να ε, καλύψουν τις προϋποθέσεις η απάντηση είναι ναι και εδώ έχουμε να κάνουμε με, ένα, με μια πράξη ισορροπίας μια προσπάθεια εξισορρόπησης ε, των πληροφοριών που απαιτούνται για να είναι ασφαλής η ε, χρήση του προϊόντος αφενός, αφετέρου προσπαθούμε και να αποφύγουμε περίτη επιβάρυνση του κλάδου. Εν προκειμένου προβλέπονται και στον κανονισμό των βιοκτώνων τον ίδιο λύσεις για ε, διάθεση στοιχείων που μπορούν να μειώσουν αντίστοιχα το κόστος, ε, αμοιβαιοποίηση δηλαδή των πληροφοριών, αλλά και η ΕΚΑ μπορεί να αναλάβει ε, ρόλο υποστήριξης προς τις υπηρεσίες, ώστε να τις διευκολύνει να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους κατά το πιο πλούστερο τρόπο. κύριε Σνάλφε θέλετε μια δεύτερη ερώτηση. Όχι, ευχαριστώ. κύριε Ντάλη, ένα λεπτό. Η πρώτη ερώτηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάνσεν. Είχαμε μια ακρόαση σήμερα, όπως σας γνωρίζετε. Η διαφάνεια είναι ένα από τα ζητήματα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και στην διαφάνεια θέλω και εγώ να τοποθετηθώ. Το λέω διότι πιστεύω ότι όλη η συζήτηση που μας έχει απασχολήσει και ως προς την ταξινόμηση της γλυφοσάτης θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η υπηρεσία σας πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στην υπόθεση αυτή και ότι θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες να έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Ένα κύριο βέβαια ελάττωμα είναι ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μελέτες που τους υποβάλλουν η παραγωγή. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες μας το είπε και ο εκπρόσωπος της ΕΚΑ, ότι δηλαδή κάνει την ε, μελέτη η ο παραγωγός προς βιομηχανίας και αυτήν την αξιολογή μετά η ΕΚΑ. Ερωτώ λοιπόν εσείς ε, τι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Κύριος Χάνσεν για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όντως, έχει ουσιώδη σημασία η διαφάνεια και για μια επιστημονική υπηρεσία όσο περισσότερο είναι η διαφάνεια τόσο το καλύτερο. Πρόκειται για μια από τις ε, βασικές αρχές και αξίες για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Ένα πρόβλημα και μόνο θα μπορούσε να ε, οδηγήσει σε κατάρρευση εργοετών. Έτσι λοιπόν χρειάζεται διαφάνεια και διαδικαστικά, αλλά και ως προς την λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων και τις βάσεις πάνω στον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία της ερώτησής σας. Η ερώτηση σας εστιάζεται στο κατά πόσον μια υπηρεσία πρέπει να κάνει την επαλήθευση με τα πειράματα ή να κάνει τα πειράματα μόνη της, τις δοκιμές, ή να στηρίζεται στα δεδομένα ε, του κλάδου ή τι θα έπρεπε να γίνεται στο μέλλον. Ο κανονισμός αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε μια εμπειρία που λέει ότι εν γέννη ο βιομηχανικός κλάδος έχει καλές επιδόσεις προς τις δοκιμές. 40-50 χρόνια με πρώτη την οδηγία για τις, επίσημε, για τις επικίνδυνες ουσίες στη δεκαετία του 70 έχουν δώσει καλά αποτελέσματα. Τούτου λεχθέντος κάθε ε, εμπειρία όπου δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα, κάθε δίδαγμα που αποκομίζουμε από τις περιστάσεις και η σημερινή σας ακρόαση είναι χαρακτηριστική, πρέπει να εξετάζεται με μεγάλη προσοχή, λεπτομέρεια και να συναγόνται τα κατάλληλα συμπεράσματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και θα είναι για την υπηρεσία να παρακολουθούμε τις συζητήσεις, τι δικές εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και σε άλλους χώρους διαλόγου ώστε να εντοπίζονται ενδεχόμενα σφάλματα ενδεχόμενες διαφορές ή στοιχεία που δεν συμπεριλήφθησαν στην τεκμηρίωση, ώστε να καλύπτονται αυτά τα κενά. Πάντως μέχρι τώρα το σύστημα έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά. Υπάρχουν σημεία ελέγχου, υπάρχει δυνατότητα και να εξασφαλιστεί η πλήρης μελέτη και να ε, ζητήσουμε από το εργαστήριο λεπτομερέστερα στοιχεία και από πλευρά της ΕΚΑ Επομένω υπάρχουν σημεία ελέγχου και μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το μέλλον την απόφαση δεν την έχει η ΕΚΑ. Τα χαιρέτησε αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν πρόκειται να προκύψουν αλλαγέ, βεβαίω και οι συνομοθέτε θα έχουν το ρόλο τους να αποφασίσουν δηλαδή αν το σύστημα όπω ισχύει τώρα, ισχύει τώρα πρέπει να αλλάξει. Η αναθεώρηση REACH, η αξιολόγηση REACH εξετάζει και την αποτελεσματικότητα της ε, εκπόνησης δεδομένων για το REACH. Και πιστεύω ότι όταν ετοιμάσει με βάση την ανακοίνωσή μας για το θέμα αυτό της προτάσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει ο διάλογος. Θέλετε να συνεχίσετε στην ίδια ερώτηση κύριε Ανταλή. Ναι, σύντομα η ΕΚΑ μπορεί να έχει ευρύτερο ρόλο η υπηρεσία Αξιολόγησης κινδύνου. Μπορεί δηλαδή να έχει την απαραίτητη υποστήριξη, ενδεχομένω και ενισχυμένο προπολογισμό για ανεξάρτητες ε, μελέτες. Κύριο Χάνσεν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν εμπόδια επιστημονικού χαρακτήρα. Είναι θέμα διοικητικό. Το να μπορεί να έχει τη διοικητική, το διοικητικό υπόβαθρο η υπηρεσία για να κάνει αυτή τη δουλειά. Τελείως επιστημονικά ή σε θέμα δεξιοτήτων, γνώσεων, αρμοδιοτήτων δεν έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως το προσωπικό πρέπει να επαντρωθεί καταλήλως. Αυτό σας το λέω διότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα εθνικό πρόγραμμα ε, δοκιμών εδώ και χρόνια με καλά αποτελέσματα. Το γνωρίζω κάπως, τον τρόπο που λειτουργεί, τους επιστήμονες που τακτικά συνεργάζονται και κάνουν δουλειά αντίστοιχη με αυτή της ε, υπηρεσίας αξιολόγησης κινδύνου. Και επομένω, αν αντεθεί ένα τέτοιο καθήκον στην ε, υπηρεσία, θα μπορούσε να το επιτέλεσε. Κύριε Γκέρλινγκ. Um, Να ευχαριστώ πολύ. Καλώ ορίσατε. Χαιρόμαστε που σα βλέπουμε. Να σας ρωτήσω κάτι για το Brexit. Υπάρχει ένα νέο πόρταλ στην ιστοσελίδα σας. Μια πύλη που καλύπτει τις επιπτώσεις του Brexit στις επιχειρήσεις αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερα για το ρίτς αυτή η προθεσμία του 18 και υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά από επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτό το θέμα. Δηλαδή, όσοι δεν είναι ταχμένοι ακόμα θα συνεχίσουν, θα συνεχίζει να ισχύει το ρίτς και δεν ξέρουμε βέβαια ποιες είναι και οι μακροχρόνιες επιπτώσει δεν περιμένω να το απαντήσετε μάλιστα το συγκεκριμένο. Αυτό που αντίθετα θέλω να ρωτήσω είναι το ποια σχέδια έχετε ως Γενικός Διευθυντής για να βοηθήσετε αυτές τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσετε ότι ανεξάρτητα πολιτικής συμφωνίας η ΕΚΑ θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται και να αποτελεσμάστε και μια ευκαιρία αυτό ίσως για την ΕΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Χάνσεν. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για το Brexit. Εμείς είμαστε σε παθητικό ρόλο, δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που αποφασίζονται στις ε, Βρυξέλλες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε ενεργητικά αντίθετα να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και γι' αυτό ακριβώς θα δείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας για αυτά τα θέματα που καλύπτουν το θέμα αυτού του διαζυγίου. Δεν προκαταλαμβάνουμε βέβαια τη νέα σχέση. Απλά και μόνο προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτό το διαζύγιο, πώς θα έχει, ώστε να υπάρχει κάποια σαφήνεια. Και χαίρομαι που η 100 έκανε αυτό, ώστε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και να προετοιμαστούν. Για το τι θα πρέπει να κάνει η ΕΚΑ και εγώ ο ίδιος οπωσδήποτε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τις διαπραγματεύσει με την κοινή διεύθυνση Grow και όλους τους άλλους εμπλεκομένους, η διεύθυνση για το περιβάλλον κλπ. Για να καταλάβουμε ακριβώς πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσει και να δούμε αν μπορούμε ήδη κάτι να εφαρμόσουμε νωρίτερα σε πρώιμη φάση. Γιατί από τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια συμφωνία όλες οι επιχειρήσεις και στην Ευρώπη των 27 και στον Μένο Βασίλειο θα αναμένουν κάποιες απαντήσεις. Αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρα. Κύριε Γκέρλινγκ, δευτερολογία. Πολύ σύντομα και ξαναλέω δεν περιμένω πολιτική απάντηση αλλά προβλέπεται η ΕΚΑ να είναι σε μια θέση όπου θα αντιμετωπίζει το ΕΒ Βασίλειο ως ε, μια χώρα σε μια δευτέρου επίπεδου κατάσταση μέλους. Δηλαδή θα συνεχίσει να πληρώνει ένα έδος ε, τέλος συμμετοχής. Ε, βλέπετε να υπάρχουν κάποια εμπόδια γι' αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση ο κύριο Χάνσεν. Εμεί βεβαίω ξαναλέω θα εφαρμόσουμε αυτά που θα αποφασιστούν στι Βρυξέλλε. Ανάλογα με τη σχέση που θα έχουμε στην συνέχεια, θα έχουμε περισσότερε ή λιγότερε δυσκολίε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αν αυτό συνεχίσει κατά κάποιο τρόπο να εφαρμόζει το ριτς Αν όμως τμήμα τη απόφαση τη συμφωνία για τη μελλοντική σχέση λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εφαρμόζει το ΡΙΤΣ και σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει και περιθώριο και χώρος για την ΕΚΑ και διασφαλίζεται η χρηματοδότηση, τότε δεν βλέπω γιατί να μην συνεχίσει να το κάνει αυτό η ΕΚΑ. Βεβαίω υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά και νομικά, προς διευκρίνηση, ώστε να είναι λειτουργική η ΕΚΑ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προβλήματα πάντως αυτού του είδου. Αυτά νομίζω θα πρέπει να ρυθμιστούν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση και ευχαρίστω να έχουμε συμβουλευτικό ρόλο κι εμεί. Ο κύριο ε, Κελπράντη, ομιλητή. Όχι, δεν είναι εδώ. Η κυρία Γιατεμάκη, έχετε το λόγο. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση. Η ΕΚΑ πώς θα μπορούσε να προωθήσει την ομαλή μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, κύριε Χάνσεν. Η ομαλή μετάβαση προς την κυκλική οικονομία αφορά τον ορισμό της ίδιας κυκλικής οικονομίας που θέλουμε. Και αφού γίνει αυτό, τότε εμεί θα τοποθετηθούμε ανάλογα με την ομαλή, λιγότερο ομαλή μετάβαση. Βέβαια, από την σκοπιά των χημικών στην κυκλική οικονομία το σημείο ισορροπία είναι τα υλικά τα οποία έχουν αξία και ανακύκλωση του, όπω όπως και τα χημικά συστατικά του, τα οποία είναι επικίνδυνα κάποια από αυτά και υπάρχουν αποδείξει ότι δεν τα θέλουμε αυτά τα χημικά πρέπει λοιπόν να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο. Αυτό είναι το ζήτημα ή το θέμα πολιτικής τέλο πάντων. Σε τελική ανάλυση, με οποιοδήποτε τρόπο και αν λειτουργήσει η ΕΚΑ, θα μπορούσε να βοηθήσει τεχνικά ώστε να κατανοήσουμε εκεί που χρησιμοποιούνται τα χημικά, εκεί δηλαδή που εισέρχονται στην οικονομία μέσω της ανακύκλωσης να το εξετάσουμε και σε επίπεδο χημικών συστατικών αλλά και σε επίπεδο προϊόντων μέσω του συστήματος ας αδειοδότησης από την ΕΚΑ. Η ΕΚΑ λοιπόν έχει συσσωρεύσει αρκετή τεχνική τεχνογνωσία για το πώς εξελίσσονται τα χημικά στην οικονομία γενικότερα και ειδικότερα στην κυκλική. Βέβαια αυτό είναι μακροπρόθεσμο, μακρόπνοο πρόγραμμα ή εγχείρημα αυτό που μπορούμε να κάνουμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την γνώση, τη βάση δεδομένων για τα χημικά, ώστε να έχουμε μια σωστή ανάπτυξη χημικών προϊόντων για την κυκλική οικονομία, ώστε να μειώνουμε τους κινδύνους από τη χρήση αυτών των υλικών. Έχουμε λοιπόν ένα διτό ρόλο να διαδραματίσουμε, να στηρίξουμε δηλαδή και να βοηθήσουμε την κατανόηση για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, αλλά και να διασφαλίσουμε το ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χημικά εκεί όπου έχουμε την επιθυμητή χρήση κυκλικής οικονομίας μαζί βεβαίως με την κατανόηση ακριβώς ε, την πλήρη των κινδύνων που επιφέρουν αυτά τα χημικά υλικά. Δευτερολογία. Ναι. Συνεχίζοντας να ρωτήσω ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο δύσκολα προβλήματα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης στην κυκλική οικονομία. Νομίζω, ο κ. Χάντσεν, από τεχνική επιστημονική σκοπιά το πιο δύσκολο ζήτημα να το απλοποιήσω για να γίνει πιο κατανοητός είναι το να αποφασίσουμε κατά πόσο θέλουμε τις ίδιες προδιαγραφές για τα ανακυκλώσιμα υλικά με αυτά που έχουμε για τα πρωτογενή υλικά ή αν αποδεχόμαστε αντίθετα εξαιρέσεις όσον αφορά το περιεχόμενο ώστε να ανακυκλώνται αυτά τελικά. Ας πούμε το κάδμιο στα πλαστικά παράθυρα PVC όπου έχουμε υψηλότερο τρεπτό όριο καδμίου τι γίνεται εκεί όμως με την ανακύκλωση. Θα έχουμε το ίδιο όπως στο καδμίου στο Πρωτογενέ με το ανακυκλώσιμο υλικό. Αυτό το θέλουμε ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Housling. Ευχαριστώ κύριε Χάνσεν που ήρθατε για το REACH. Το R σημαίνει registration, δηλαδή καταχώρηση ουσιών αλλά και εκεί ξεκινούν και τα προβλήματα. Δέκα χρόνια που λειτουργεί το REACH, μόνο 16% των καταχωριστικών ουσιών, 60% των καταχωριστικών ουσιών δεν αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι μπορεί στο μέλλον να ε, στοιχειοθετούνται οι φάκελοι για την καταχώρηση και επίσης πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε προστασία τη δημόσια υγεία και του περιβάλλοντος από επικίνδυνε ουσίες. Γίνονται αδειοδοτήσει για ουσίες οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί κατά τρόπο αξιόπιστο. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο των αδειοδοτήσεων ώστε να βρεθεί η εναλλακτική στην ουσία που μπορεί να είναι επικίνδυνη και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Thank you. Thank you very... Ευχαριστώ. Το ερώτημά σας νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί σε δύο σκέλη. Πρέπει δηλαδή να εργαστούμε ουσιαστικά πάνω σε δύο άξονες. Αυτό εννοώ. Αλλά πρώτα απαντήσω, θέλω να πω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η ΕΚΑ προσπαθεί να λειτουργήσει σωστά ο κανονισμός σε και να έχει αποτέλεσμα. Και συμμερίζομαι την εντύπωση που έχετε για το πώς αποδίδευσε ο κανονισμός αλλά νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Το επόμενο βήμα, και εδώ έρχομαι στο ερώτημά σας, πώς θα είμαστε πιο αποδοτικοί για να έχουμε καλύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων και περισσότερη δουλειά να επιτελείται στο επίπεδο ΕΚ. Δύο είναι τα σκέλη, δύο είναι άξονες. Ο πρώτος είναι ότι μετά από 10 χρόνια εφαρμογής του REACH, η αρχίζει πλέον να να σωρεύει εμπειρία και γνώση για τα χημικά, κάτι το οποίο επεμβαίνει το εκάστοτε χημικό προϊόν, την εκάστοτε απόφαση. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να προωθήσουμε τη γνώση την επιστημονική για τις χημικές ουσίες και να την αξιοποιήσουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, καταχώρηση, αξιολόγηση, περιορισμοί, αδειοδοτήσεις κτλ ώστε η λήψη αποφάσεων να γίνεται ταχύτερα και καλύτερα. Υπάρχουν όμως ε, και κέρδη γενικά ε, ως προς την αποδοτικότητα. Τα συζητάμε σε επιτροπές και με το προσωπικό. Δηλαδή, κάθε φορά που λαμβάνεται μια απόφαση πρέπει να αντλήσει και ένα δίδαγμα από αυτή την απόφαση. Δέκα χρόνια μετά λοιπόν ένα καλό το χρονικό πλέον διάστημα που έχει έρθει για να δούμε τι έχουμε διδαχθεί. Πού μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο γρήγορα. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να απαντήσω άλλα 24 λεπτά για το θέμα αυτό. Πώς περάσαμε στο ρίτσα από την προηγούμενη νομοθεσία. Κάναμε πολλή δουλειά θεωρητική, προβληματιστήκαμε, αναστοχαστήκαμε και μετά τα 10 χρόνια έχουμε και την αξιολόγηση του Ριτς από την Κομισιόν, αλλά και ΕΚΑ μπορεί να κάνει μια πιο τεχνική επιστημονική αξιολόγηση, ώστε να έχουμε περισσότερη αποδοτικότητα και ταχύτερη λήψη αποφάσεων, κάτι που θα ωφελήσει εν τέλει τους πολίτες. Ευχαριστώ. Έχετε να κάνετε και μια δεύτερη ερώτηση. Ανήκουν στις προτεραιότητές σας, τέλο πάντων ποιες είναι οι πρώτες σας τρεις προτεραιότητες, καλύτερα να μου πείτε. Απάντηση. Μ, ναι. Υπάρχουν πολλές προτεραιότητε το να έχουμε αποδοτικότητα πράγματι ως οργανισμός είναι μία προτεραιότητα, όχι μόνο για να έχουμε την πλήρη εφαρμογή των τεσσάρων και συντόμως πέντε νομοθετημάτων στον τομέα μας, αλλά για να δείξουμε ότι η ΕΚΑ μπορεί να φιλοξενήσει εντός εισαγωγικών και άλλα νομοθετήματα για τα χημικά. Αυτή είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Οι άλλε πολύ σημαντικέ προτεραιότητε, μάλλον η άλλη πολύ σημαντική προτεραιότητα είναι σε πέντε χρόνια από τώρα η ΕΚΑ να μπορεί να αξιοποιείται και να χρησιμοποιείται πολύ καλύτερα ω η κατεξοχήν ε, οργάνωση που, που έχει τη γνώση και την τεχνογνωσία στο θέμα σε Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε ο γύρος ε, τα απαντήσεων από του συντονιστέ ε, και περνάμε στο δεύτερο γύρο. Δεν έχω βέβαια ούτε και εδώ ένα μακρύ κατάλογο, οπότε αν θέλει οποιοδήποτε άλλο ε, μπορεί να σηκώσει το χέρι. Κυρία Κάντεμπαχ είναι η πρώτη στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάνσεν που είστε εδώ και για την διάθεσή σας να απαντήσετε. Ήδη απαντήθηκαν κάποια από τα ερωτήματά μου. Δύο σύντομα σχόλια μου επιτρέπετε. Το ερώτημά μου είναι εσεί προσωπικά πώ αντιμετωπίσετε τι εκθέσει του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ε, την απαλλαγή βαρών και την ε, απαλλαγή. Υπάρχουν κάποιες ε, εκθέσεις Ελπίζω να λαμβάνετε υπόψη τις συστάσεις παραδείγματο χάρη ό,τι αφορά την κατάρτιση δικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Και το δεύτερο, επαναρχόμενο σε ένα ερώτημα που ετέθη πριν, τη δυνατότητα ή το καθήκον της ΕΚΑ ε, να έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο, υποστηρικτικό ρόλο σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία και το αναφέρω σε σχέση με τις χημικές ουσίες. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά ως προς την κυκλική οικονομία στον τομέα αυτό. Κύριε Χάνσερ, απάντησε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πολύ διαφορετικά ερωτήματα. Αλλά ναι, όπως πολύ σωστά προβλέπετε, Φυσικά και λαμβάνω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ε, ε, τις θέσεις του Κοινοβουλίου και τα όσα ε, προ στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κύκλου. Πάντοτε, σε όλη μου τη σταδιοδρομία στις Βρυξέλλες, παρακολουθούσα τα θέματα του σύνεγγις και παρακολουθώ και το δημοσιονομικό κύκλο και το πώς λειτουργεί και είναι ικανοποιητικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί όπως φαίνεται και βέβαια οτιδήποτε προκύπτει συζητήσει ε, αναφέρεται, υποβάλλεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης γίνονται προτάσεις από τη Γραμματεία, η ανάληψη δράσης ε, ως απάντηση σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη κριτική ή σχόλιο. Και μετά όλα αυτά συζητούνται στο σχέδιο δράσης ε, σχεδιασμού. Και συζητείται και εγκρίνεται στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τελευταία 10 χρόνια η σχολιο και μετα ολα αυτα συζητουνται στο σχεδιο δρασης σχεδιασμου και συζητειται και εγκρινεται στο επιπεδο του διοικητικου συμβουλιου τα τελευταια 10 χρονια εμπειρια μα δείχνει ότι αυτό ο κύκλος συνεχού βελτίωση ότι δηλαδή αναλαμβάνει ουσιαστικά την ευθύνη το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, φαίνεται να αποδίδει τρόπο εργασία. Γιατί όλο και λιγότερα προβλήματα ανακαλύψει τη δικασία απαλλαγή η ε, Επιτροπή Προπολογισμού. Α, και επειδή υπήρχε και το δεύτερο ερώτημα για την κυκλική οικονομία, ε, πολύ γρήγορα να πω ότι ΕΚΑ έχει τι δικέ τη αρμοδιότητε ε, και ο στόχο τη είναι να βοηθήσει τους ε, θεσμούς να εφαρμόσουν δεσμέτρων για την κυκλική οικονομία με όποιον τρόπο αυτό αποφασιστεί ε, ότι πρέπει να γίνει από πλευρά ΣΕΚ. Και η σαυσάρμοντα της ΕΚΑ είναι να καταλάβει την τοξικότητα μεν, αλλά και την χρήση των χημικών σε όλο τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή και τη διάθεση και την ανάκτηση και την ανακύκλωση. Άρα η αρμοδιότητά της είναι σημαντική, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που θα ακολουθηθεί, θα αποφασιστεί από πολιτικής πλευράς ε, για την κυκλική οικονομία. Είτε πρόκειται για ίση αντισώτη ε, μεταχείριση ανακύκλωσης ανακυκλωμένων υλικών και πρωτογενών υλικών, είτε υπάρξει η δυνατότητα εξαίρεσης για κάποια δευτερογενή υλικά. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστούμε τον κύριο Χάνσεν που είναι εδώ. Ε, προσωπικά ένα σχόλιο και μετά ένα ερώτημα. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιληφθούμε τη σημασία τη ύπαρξη ενό θεσμού όπω η ΕΚΑ. Ο στόχο σα είναι να αξιολογείτε όλε τι χημικέ ουσίε που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βλέπετε αν έχουν τι ιδιότητε ε, που λένε ότι έχουν ή όχι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτόν τον οργανισμό με τόσο καλούς εμπειρογνώμονες που εργάζεται με τόσο επιστημονικό τρόπο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πέσουμε στην παγίδα του να έχουμε πολιτικές συζητήσεις και να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Το ερώτημά μου σχετίζεται λίγο με το όσα έλεγε η κυρία Ντάλη πιο πριν για τη διαφάνεια. Φυσικά και πρέπει η ΕΚΑ να είναι ένας αξιόπιστος ε, συνομιλητής και η Επιτροπή Εξόλυξης Κινδύνου είναι πολύ σημαντική. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να έχετε τις δυνατότητες να φέρετε σε πέρα στο έργο σας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάτι σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που λαμβάνετε. Σε ποιο ύψος είναι. Και τι γίνεται και με τον Brexit στη συνέχεια. Νιώθω ότι έχετε αρκετή χρηματοδότηση και για το μέλλον ενώπιση του Brexit. Πώ μπορούμε εμεί να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση και ποιο είναι ο δικό σα ρόλο. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Δύο τμήματα βλέπω στην ερώτησή σα το γενικό θέμα τη χρηματοδότηση και εξασφάλιση τη δουλειά, τη ΕΚΑ και ιδιαιτερότητε. κάθε πρόσθετη δαπάνη που μπορεί να προκύψει, κόστο που μπορεί να προκύψει λόγω του Brexit. Ο ρόλο μου και μια από τι κύριε λειτουργίε μου είναι να εξασφαλίζω ότι θα υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση ή ότι θα, είναι, θα καθίστανται γνωστά ε, όποια ελλείμματα στη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην, ε, μέσα στον κύκλο της ε, ε, κατάρτισης και εκτέλεσης του προπολογισμού. Και πέραν αυτού, δουλειά μου θα είναι επίσης να κοιτώ και μακροπρόθεσμα τι άλλο μπορεί να γίνει για να ε, καλυφθούν οι ανάγκες ένωση σε θέματα προστασίας ε, στα χημικά και να επιτελείται το έργο της υπηρεσίας επαρκώς. Εδώ υπάρχει σημαντικό δυναμικό, ε, πιστεύω, εάν βέβαια υπάρχει και πολιτική βούληση για αξιοποίηση των γνώσεων που έχει αναπτύξει η υπηρεσία της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων που έχει η υπηρεσία και, η, και το προσωπικό της ώστε να κάνει τη δουλειά της καλύτερα. Στο κόστος που να προκύψει από το Brexit από την προοπτική των Βρυξελών μπορώ να πω ότι α, δεν θα είναι και τόσο μεγάλο, αλλά αυτό χωρίς να έχω μιλήσει με την υπηρεσία. Και με βέβαιος ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο ε, περίπλοκη από ό,τι μπορεί να δει κανείς από τις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ λοιπόν να δώσω απάντηση τώρα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το κοιτάξουμε. Δεν θα είναι το απλούστερο πρόβλημα αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει νέα συμφωνία και μόνο διαζύγιο, αυτό δεν ισοδυναμεί με το να κόψει κανείς την τηλεφωνική γραμμή προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλά περισσότερα πράγματα θα γίνουν για να πραγματοποιηθεί ε, ομαλά η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από το ρυθμιστικό σύστημα. αλλά το τι ακριβώς κόστος θα φέρει αυτό δεν το ξέρουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Ντός. Δεν ήξερα ότι θα φτάνατε τόσο γρήγορα σε μένα. Ευχαριστώ που έχετε απαντήσει αυτέ τις ερωτήσεις μέχρι τώρα. Θα διατυπώσω άλλη μία για τον Brexit και ζητώ συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνετε ότι με απασχολεί πολύ. Είμαστε λοιπόν σε ένα στάδιο που πια πρέπει να προχωρήσουμε εφόσον οι συνθήκες και οι πολιτικοί εγωισμοί στη Βρετανία το επιτρέψουν και ένα πράγμα που μου φαίνεται πιο εντυπωσιακό στους εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε τομέα είναι ότι λένε πάντοτε ότι θέλουν τη σύγκληση τη ρυθμιστική με τον ευρωπαϊκό χώρο. Ε, πάνω απ' όλα γιατί είναι αυτές οι αγορές τις οποίες δραστηριοποιούνται. Ξέρω ότι θα μου δώσετε κάποια, ας το πω έτσι, διπλωματική απάντηση, αλλά τι συνέπειες θα φέρει στο εμπόριο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο το ε, ενδεχόμενο να υιοθετήσει δικό του ρυθμιστικό καθεστώς το Ηνωμένο Βασίλειο άπαξ και ολοκληρωθεί το Brexit, γιατί αυτό προτείνουν ορισμένοι που υποστηρίζουν την ιδέα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένες ιδέες για το τι είδους συνέπειες μπορεί να φέρει στο εμπόριο, πιθανές συνέπειες μεταξύ των δύο αυτών ε, ε χώρων των εμπορικών μπορεί να φέρει. Να και που έχετε και ερώτηση για το εμπόριο, λέει η κυρία Βαλιάν, ο κύριος Χάνσεν. Ας πάω πίσω ένα βήμα πριν να αρχίσω με αυτή τη φράση. Το ρίτς έχει ένα κόστος και τα ωφέλη του έρχονται μετά. Υπάρχει το κόστος στην ε, καταχώρηση, στην δοκιμή των χημικών, στην κοινοποίηση των δεδομένων μεταξύ όλων των εισαγωγείων ή παραγωγών, της ίδιας ουσίας, κόστος από την αξιολόγηση κινδύνου, κόστος από τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που εξασφαλίζουν ότι η ουσία είναι υπό έλεγχο σε όλη τη διαδικασία, σε όλη την αλυσίδα προμήθεια. Σα το λέω ε, αναλυτικά γιατί είναι σημαντικό το εμπροστοβαρέ κόστο. Τα ωφέλη έρχονται εκ των υστέρων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση και με το προθεσμίο του 2018 γιατί οι βρετανικέ επιχειρήσει έω το Μάιο, στι 31 Μαΐου του 2018 θα έχουν ε, επενδύσει, θα έχουν υποστεί δηλαδή αυτό το κόστο. Τα ωφέλη όμω θα έρθουν μετά με μια διαφανή και ομοιογενή αγορά, όπου όποιος έχει κάνει καλά τη δουλειά του θα δει και την ανταμοιβή. Βέβαια μετά, εάν πραγματοποιηθεί ένα διαζύγιο που δεν θα έχει άλλη συνέχεια, άλλη συμφωνία δηλαδή που θα το ακολουθεί, τα ωφέλη που θα μπορούσε κανείς να αποκομίσει όταν θα είναι η Ευρώπη μόνο το 27 δεν θα έρθουν. Ε, ας δούμε λοιπόν ποιε είναι οι εταιρείε οι οποίες ε, έχουν έδρα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλές είναι αυτές που ονομάζονται omni-representatives, δηλαδή γενικοί ε, αντιπρόσωποι, δηλαδή εισαγωγή για όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο, και έχουν βέβαια και την προσβασιμότητα, τη διευκόλυνση προσβασιμότητα στις εθνικές αρχές που θα τους αδειοδοτήσουν. Αυτές έχουν κάνει μια αξιολόγηση αυτές οι εταιρείε και έχουν δει ότι για να αποκομίσουν ωφέλη ενδεχομένως να χρειαστεί να μετατοπιστούν. Βεβαίως υπάρχει το ζήτημα και των Βρετανών, καθαρά Βρετανών ε, κατασκευαστών σημαντικό πάλι νούμερο ε, επιχειρήσεων, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, όπου πάλι αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τους κανόνες του, θα, θα εφαρμόζονται οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και ως εκ τούτου θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές εταιρείε αυτές στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα έχουν ήδη κάνει την επένδυση. Ευχαριστώ κύριος Μπράνεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Λυπούμε που δεν είναι πιο πολλοί οι βουλευτές. Αλλά είχαμε και 3,5 ώρες συζήτηση για τη γλυφοσάτη σήμερα το πρωί. Δεν κάνει καλό στην υγεία των ευρωβουλευτών από ό,τι φαίνεται αυτό. Με ενδιαφέρον σημειώνω ότι οι σοσιαλιστέ έχουν καλύτερη ανθεκτικότητα στην έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες από ότι άλλε πολιτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου. Αντίστοιχη με την ερώτηση της Τζούλιαν και του ΣΕΠ, καθώς είμαι και εγώ Βρετανός Ευρωβουλευτής, θα είναι και δική μου ερώτηση. Ε, ως επιστήμονας ξέρω ότι δεν θα κάνετε τυχαίες υποθέσεις, αλλά και χωρίς να θέλω να σας τραβήξω σε μια ε, υπόθεση εναλλακτική, Ποιε θα ήταν οι καλύτερες, ε, τα καλύτερα ενδεχόμενα για την εξέλιξη του Brexit, γιατί τα χειρότερα σενάρια μπορούμε ξέροντάς τα να τα αποτρέψουμε ενδεχομένω. Παρακαλώ. Χειρότερα σενάρια λοιπόν, οι χειρότερες εκδοχές, τα πιο ακραία σενάρια που θα μπορούσα ε, εκ του προχείρου να σκεφτώ, θα ήταν διαζύγιο χωρίς διευθέτηση, χωρίς συμφωνία δηλαδή για το πώς οι βρετανικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να διαφυλάξουν την επένδυσή τους σε σχέση με την Ευρώπη των 27, όπου τα προβλήματα αφενός θα είναι για τις, 27, ε, για τις εταιρείες των 27 της Ευρώπης, όταν δεν έχουν αποφασίσει οι Βρετανικές εταιρείες να επανεγκατασταθούν ή να ε, εγκαθιδρύσουν ε, θηγατρική ή υποκατάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Άρα οι επιχειρήσεις αυτές των 27 εναπομεινασών χωρών θα έχουν ε, πάλι απώλεια των επενδύσεών τους. Αν και όπως είπα θεωρώ ότι θα είναι πολλές αυτές οι επιχειρήσεις που από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ε, φτιάξουν υποκαταστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Το αντίστροφο όμως είναι πιο πιθανό, δηλαδή να μην είναι στη διάθεση του Ηνωμένου Βασιλείου πλέον ούτε της βιομηχανίας ε, αλλά ούτε και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τα δεδομένα και τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις των 27 ε, κρατών μελών που θα έχουν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο σε ένα διαζύγιο χωρίς συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Ροστέτ. Λυπάμαι που καθυστέρησα, αλλού ήμουνα και σας άκουσα. Άκουσα και τις καλές ερωτήσεις των συναδέλφων για τις επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit. Επ' αυτή την προοπτική, γνωρίζοντα ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία και πάμε προς σκληρό Brexit, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τότε η αντίδραση του Νέου Βασιλείου θα ήταν να πει ότι εγώ θα μειώσω φόρους για να έρθουν σε εμά όσοι θέλουν να επενδύσουν, αν το πει αυτό η Ένωση, η Βρετανία θα πει εντάξει δεν πειράζει, θα κάνουμε με πολύ διαφορετικά. Αυτός είναι ένα κίνδυνο. Γιατί σημαίνει αρχικά ότι θα έχουμε ύφεση στο Νέο Βασίλειο που μπορεί ενδεχομένω να πάει και αλλού μου στο Νέο Βασίλειο, να βρει αλλού, να αναζητήσει αλλού εταίρου, είπα και λοιπά. Και η ύφεση στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει ύφεση και στην Ένωση αφορά και τις δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν μας αποδεικνύει ότι δεν θέλουμε σκληρό Brexit. Οι επιχειρήσεις όμως οι χημικές δεν χρειάζεται να τηρήσουν τις δεσμεύσεις μας και τους περιορισμούς μας. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα γιατί αποτελεί μια υποχώρηση. Εσείς πώς το βλέπετε. Εσείς λέτε ότι να αποδείξουμε ότι αυτά που κάναμε στο ρίτς ε, ας πούμε, όντως είναι μια σημαντική πρόοδος και πράγματι έτσι είναι για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, όμως έχει και κόστος. Το οποίο, το οποίο όμως το ωφέλη στη συνέχεια αργότερα. Εντάξει, αλλά αν όμως η εταίροι μας αυτοί αποφασίσουν να μην τηρήσουν τίποτα και να πάρουν οικονομικά μέτρα τα οποία θα κάνουν δύσκολη θα ισχυρένουμε από τον ανταγωνισμό με την Ένωση, τότε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εγώ πραγματικά να σου πω ανησυχώ για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω σε ένα τμήμα της ερώτησης, γιατί πολλά από αυτά που είπατε είναι εκτός δικιάς μου αρμοδιότητας. Και δεν ξέρω τι θα κάνει το Βασίλειο ακριβώς για να ζητήσει αλλού εκτήματα ή όχι. Δεν έχω λοιπόν αρμοδιότητα να πω κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό μπορώ να πω ξεκάθαρα τώρα και να επαναλάβω με άλλα λόγια είναι ότι οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έκαναν επενδύσεις, έχουν την καταγραφή τους στο Μητρό, έχουν πρόσβαση, έχουν κάνει εξολογήση κινδύνου, έχουν εφαρμόσει μέτρα για να διασφαλίσουν την ε, σωστή χειραγώρηση και χρήση. Αυτή η επένδυση δεν αφορά μόνο την υγεία και το περιβάλλον, αλλά αφορά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στις διάφορες αλυσίδες και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν υγείας και περιβάλλοντος, είναι εμφανώς, αλλά έχει και προεκτάσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι προηγουμένω ανεξάρτητα του συστήματος που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το Ενωμένο Βασίλειο, αυτό η δουλειά του Ενωμένου Βασιλείου και αποτέλεσμα τη διαπραγμάτευση. Όμω, παραμένει το γεγονό ότι οι επενδύσει που έχουν γίνει έχουν γίνει. Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Οπότε, οι... τα προποτούμενα προδιαγραφέ REACH τηρούνται από τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όσον όπως λέξα, και η έκθεση πούμε, για τα δεδομένα αυτά της μεταποίησης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, να ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάνθεν στην τελική του δήλωση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω μια πολύ σύντομη δήλωση. Από τη μια χαίρομαι που δεν υπάρχουν περισσότεροι βουλευτές, οπότε σταμάτησε το μαρτύριό μου, ήταν πιο περιορισμένο. Αλλά είδατε από τα προκατακτικά μου σχόλια κάποιοι από εσά που είσαστε ενεργοί σε αυτό το ε, τομέα, έχετε και τεχνογνωσία, έχετε γνώσεις. Προσλέπω να συνεργαστούμε μαζί τα επόμενα πέντε χρόνια, ώστε να προωθήσουμε και βοηθήσουμε στη δουλειά μας και την εφαρμογή, αλλά και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων που έχει η ΕΚΑ προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι η σύντομη μου δήλωση και σας ξανά ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε και κυρίε και κύριοι βουλευτέ για τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω οι απαντήσεις μου να συνέβαλαν στο να με δείτε υποθετικό φως τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Χάντσεν. As uh, Όπως είπαμε στην αρχή, ξεκινήσαμε κατευθείαν με την ανταλλαγή απόψεων, αλλά τώρα επανέρχομαι στο αρχικό σχέδιο ως είχε της μερισίας. Την είδατε. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις ή να την θεωρήσουμε εγκεκριμένη. Και μετά από έτοιμα της κυρίας Σεύκοβιτς. Είχαμε ένα μια ανταλλαγή απόψεων την οποία αναβάλουμε 27 του Νοέμβρη και το τελευταίο σημείο της ημερήσιας θα συζητηθεί αργότερα. Θα το δούμε μετά τις ψηφοφορίες. Αυτές τις δύο ανακοινώσεις είχα να σας κάνω σε σχέση με τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε ένα workshop που προεδρεύουν Καπασόν και Πέτερλινγκ στις 16 του Οκτώβρη σε σχέση με συμπληρωματικές και εναλλακτικέ θεραπείες για τους ασθενείς σήμερα και αύριο. Αρχίζει στις 4 και σας καλώ να συμμετάσχετε θα έχουμε επίσης μια έκτακτη συνάντηση επιτροπής μας στο Στρασβούργο τη Δευτέρα. 7.30. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης για τις ανανεώσιμες. Έχετε λάβει τους ηλεκτρονικούς φακέλους και θα έχουμε και δερμηνία. Επίσης, ηλεκτρονικά λάβατε και τις συστάσεις των συντονιστών και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της μέρας, τι θεωρούμε εγκεκριμένε. Τώρα, πάμε στο σημείο 6. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και την εααταφ σχετικά με τους γενικά τροπομένους οργανισμούς για τα κριτήρια για την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου να επιθυμίσω ότι μετά από αίτημα των πρασίνων αποφάσισαν οι συντανιστέ να γίνει αυτή η ανταλλαγή, ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις, δηλαδή σήμερα. Και χωρίς να καθυστερήσω άλλο, θα δώσω το λόγο στην Εύσα και την Επιτροπή για 15 περίπου λεφτά. Σαμπινούλη και από την Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για, αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπως ξέρετε πολλοί από εσά, στο τέλος της εβδομάδας θα υποβάλει η Κομισιόν στη Ρυθμιστική Επιτροπή μια ανταλλαγή απόψεων και ένα σχέδιο γνωμοδότησης για μια οδηγία της Κομισιόν που τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας 2018. Βασιζόμενοι στις κατευθυντήριες γραμμές της ε, τωρινές της ΕΦΣΑ όσον αφορά τα γενικά τροπημένα γενικά οργανισμούς, ιδιαίτερα τα φυτά τα που είναι γενικά τροπημένα προς καλλιέργεια στην Ένωση. Αυτό λοιπόν το σχέδιο οδηγίας συντάχθηκε σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας opt-out και είναι σύμφωνη με τα αντίστοιχα άρθρα της οδηγίας που μιλούν για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο. Να σας διαβεβαιώσω ότι είχαμε εκτεταμένες συζητήσει με την ΕΦΣΑ αφενός για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κύρια στοιχεία του καθοηγητικού εγγράφου θα περιληφθούν στο σχέδιο του κειμένου μας και αφετέρου είχαμε ευρύ συζητήσει τεχνικές με τις χώρες μέλη για το σχέδιο της οδηγίας που διευκρινίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις διατάξεις. Να πω ότι αυτό το κείμενο περιλαμβάνει και μια τεχνική ενημέρωση και ε, που δεν, δεν επιφέρει μια αλλαγή πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Ιδιαίτερα μιας και μιλάμε ε, για τροποποιήσεις κάποιων παρατημάτων της οδηγίας. Θεωρούμε ότι καταρχάς με αυτές τις τροποποιήσεις στηρούμε τη νομική μας υποχρέωση που θα έπρεπε να είχαμε υλοποιήσει μέχρι το Απρίλη και κυρίως να ενισχύσουμε κάποια θέματα κάποια σημεία δηλαδή να μειώσουμε κάποιε αβεβαιότητε όσον αφορά τωρινή μεθοδολογία αλλά και σε θέματα όπως υποβολή των δεδομένων να ακολουθήσουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Θα σκεγγραφίζω τις πιο κύριες αλλαγές. Όπως σας είπα, μα ζητήθηκε να δουλέψουμε βάση του τωρινού εγγράφου τη γραμμών της ΕΦΣΑ και αυτό που κάναμε είναι να ενσωματώσουμε τα κύρια στοιχεία αυτού του εγγράφου καθοδήγησης, δηλαδή η μεθολογία έξι βημάτων για την ε, αποτίμηση του κινδύνου των γενικά οργανισμών. και λεπτομερέστερα για τα φυτά, τα γενικά τροπεμένα και τα συμπεράσματα που αφορούν συγκεκριμένου και αντίστοιχους τομεί κινδύνου. Εξετάσαμε τη μεθοδολογία λοιπόν και με την ευκαιρία εξετάσαμε και κάποια πιο οριζόντια ζητήματα όπως οι μακροχρόνιες παρενέργειες, ποιότητα δηλαδή των δεδομένων που υποβάλλονται, και άλλα αντίστοιχα στοιχεία. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας ότι αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές της ΕΦΣΑ αφορούν τη θέση στο εμπόριο αυτών των φυτών τη στιγμή που οι περισσότερες διατάξεις αφορούν όλα, όλους τους γενικούς τροπομινούς οργανισμούς και κατά, κατά την παραγωγή τους και κατά τη διαθέση στο εμπόριο. Στα παραρτήματα είδαμε ότι κάποιες προαπαιτήσεις για τα δεδομένα δεν σχετίζονται μεταξύ και κίνδυνο όσον αφορά τη θέση του εμπόριου αυτών των φυτών και γι' αυτό ακριβώ θα θέλαμε να υπάρχει ευθυγράμμιση με την διαδικασία αδειοδότηση των φυτών αυτών, ώστε οι απαιτήσει των δεδομένων να απαριθμώνται στην, ε, με την ίδια σειρά και να χρησιμοποιείται η ορολογία. Ήδη καταλαβαίνετε από αυτά ότι ήδη είχαμε μια αρκετά τεχνική δουλειά και μια αρκετά τεχνική διαδικασία ενημέρωσης. Δεχτήκαμε ερωτήσεις παλαιότερα σε σχέση με τα εκτιμώντας ιδιαίτερα το 9 και μας ζητήθηκε να διευκρινίσουμε κάποια θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά την διάδραση μεταξύ νομοθεσίας που αφορά τα γάματα όμικρον και τα ζανιοκτώνα, τα αυτοφάρμακα. Και πάλι δεν θεωρούμε ότι υπάρχει εδώ κάποια αλλαγή πολιτικής, απλά και μόνο επιφέρουμε κάποιες διευκρινήσεις. Κατά την άποψή μας, είναι σημαντικό να διευκρινίζεται σε αυτό το ζήτημα, στην τροποποίηση αυτής της οδηγίας και όσον αφορά τη νομική σκοπιά, αλλά και την επιστημονική. Από την νομική σκοπιά, οι άδειε για τους γάμματα φωμικρών δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα σε σχέση με τη χρήση των φυτοφαρμάκων, επειδή αυτά τα μέτρα αφορούν μόνο την νομική βάση της νομοθεσίας που συνοδεύει τα φυτοφάρμακα. Και από επιστημονική σκοπιά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πρακτική εμπειρία όσον αφορά την αντοχή στα ζωνιοκτώνα σε σχέση με την καλλιέργεια. Οπότε ε, δεν έχουμε κάποια μακροχρόνια δεδομένα να λάβουμε υπόψη μας. Επίσης ε, δεν υπάρχει αδειοδότηση, αδειοδότηση χρήσης κάποιων προϊόντων προστασία όσον αφορά την ε, χρήση αυτών των ε, γαμματάφ όμικρον και αν υπήρχε θα έπρεπε να διοδετηθεί υπό, την, ε, υπό τις διατάξεις και τα προπόμενα της οδηγίας για τα φυτοφάρμακα. Να σας πω και δύο λόγια σε σχέση με την αδειοδότηση των προϊόντων προστασίας των φυτών θα αποφεληθούμε τις της ΕΦΣΑ όσον αφορά την τεχνική της γνώση και την τεχνογνωσία Έχουμε όμως μια διαδικασία αδειοδότηση όπου το ενεργό συστατικό αδειοδοτείται σε επίπεδο ένωσης, προβάθμια και μετά σε δεύτερο στάδιο αφορά τα προϊόντα φυτών και μετά τις χρήση, τη χρήση του στις χώρες. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι η αποξελόγηση κινδύνου εκ μέρους των χωρών είναι υποχρεωτική όσον αφορά όλες τις χρήσεις και αυτό σημαίνει επίσης ότι οι αλλαγές όσον αφορά την χρήση μετά από την ε, εισαγωγή αυτών των ε, γαμματαφόμικρων οι χώρες μέλη θα πρέπει να κάνουν μια νέα αξιολόγηση κινδύνου. Για τα προϊόντα προστασία ε, φυτών θα πρέπει να εξεταστούν επίση και οι περιβαλλοντικέ ιδιαιτερότητε των χωρών μελών, όπω α πούμε κλιματικέ συνθήκε κλπ. Και οι χώρε μέλη επίση θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπιση τα οποία θα προσυδειάζουν στην κατάσταση αυτή στην κατάστασή τους. Οπότε, για να είμαστε ξεκάθαροι, στην πράξη μιλάμε για μια διαδικασία σε δύο βήματα, όπου αφενός η πιθανή αντιδότηση του γαματαφόμικρου θα αξιολογείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ΕΦΣΑ και σε τελική ανάλυση ε, το φυτό ή το προϊόν που θα διδοτείτε θα διαχωρίζεται από την χρήση των φυτοφαρμάκων ω προϊόν ως γαματαφόμικρον και θα συνοδεύεται από αξιολόγηση κινδύνων, δηλαδή από την χώρα η οποία θα επιτρέπει την καλλιέργεια αυτού του γαματαφόμικρον και θα πρέπει να λαμβάνει βεβαίως υπόψη τη τι της συνθήκε στην κάθε χώρα μέλο. Ενημερωτικά τώρα, να σα πω για κάποια άλλα διαδικαστικά ζητήματα. Όπως σας είπα, είχαμε εκτενείς συζητήσεις με την ΕΦΣΑ και με τις χώρες μέλη και κοινοποιήσαμε στο SPS και στο TPT τα αποτελέσματα και η πρόταση αυτή ήταν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης για εβδομάδες όπου δεχτήκαμε κάποιες παρατηρήσεις από τους ε, ενδιαφερόμενους και τα σχόλια που λάβαμε αναλύθηκαν και λήφθηκαν υπόψη στο μέτρο του δυνατού όταν ενημερώσαμε το σχέδιο της οδηγίας. Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι οι αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας στήριχθηκαν πλήρως, ότι όλα τα βήματα της διαδικασίας που προκαθόρισαν οι νομοθέτες ε, για τους γάμματα φωμικρών έχουν ακολουθηθεί και Νομίζω ότι επίσης δεν ε, υπερβήκαμε την εντολή μας και κυρίως νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε στην ε, νομική μας υποχρέωση που μας επέβαλε ο σύνομαθέτης μέσω δηλαδή της ε, προσαρμογής στην τεχνική εξέλιξη, τεχνικές εξελίξεις. Θα ενισχυθεί λοιπόν η αξιολόγηση αυτών των γάμματα φόμικρων με αυτά τα μέτρα, μειώνοντας ακριβώς τις ανασφάλειες και ενισχύοντας τη μεθοδολογία. Και όπως σας είπα, η υποβολή των δεδομένων με αυτό το μέτρο θα ακολουθεί το βήμα των, των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ταραζόνα. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Από την προοπτική της ΕΦΣΑ φυσικά δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε εξέταση κινδύνου στην περίπτωση αυτή και η περιβαλλοντική εκτίμηση και για τα φυτοφάρμακα και για τα ζανιοκτώνα είναι κάτι πολύ σημαντική και βέβαια για τα ζανιοκτώνα αυτό πρέπει να γίνει είναι να αξιολογηθεί η δραστική ουσία αφενός και είναι ευθύνη των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ ε, πριν να διοδοτήσουν οποιοδήποτε φυτοφάρμακο. Η μεθοδολογία φυσικά και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Υπάρχει ε, η καθοδήγηση, υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές από την ΕΦΣΑ. Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση φυτοφαρμάκου υπάρχουν διάφορες ε, μελέτες και διάφορες συστάσεις από διάφορους φορείς για την περιβαλλοντική εκτίμηση αντικτύπου και βέβαια μεταξύ των ευθυνών μας και των υποχρεώσεων μας είναι να δίνουμε γνωμοδοτήσεις. Έχουμε την Επιστημονική Επιτροπή τη ΕΦΣΑ που καλύπτει όλους τους τομείς και σε περιλαμβάνεται εκεί και η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικού αντικτύπου και η μελέτη των ζανιοκτώνων και των φυτοφαρμακευτών τα ζανιοκτώνα. Υπάρχει εναρμόνιση. Οι διευθυντή εξόρου κινδύνου θα κάνουν βέβαια, θα λάβουν τι αποφάσει βάσει τη τη ΕΦΣΑ. Πάντως έχουν προχωρήσει εργασίες, έχουμε βέβαια απόφαση των νομοθετών, ε, δεν είναι θέμα της ΕΦΣΑ. Αλλά αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι με αυτό το σύστημα θα έχουμε την αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της δραστικής ουσίας καταρχάς και μελέτη όλων των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων. Και έπειτα αξιολογείται κάθε φυτό ξεχωριστά και κάθε χρήση του. για να υπάρχει ώστε να το μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, απλά επιβεβαιώνουμε ότι σε ό,τι αφορά τα, τη χρήση των ζενεπτώνων σε καλλιέργειες σε γάμματα φωμικρόνα, ορίζεται πολύ καλά σε αυτά που προτείνονται και νομίζουμε ότι θα καθιερώσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστούμε. Ποιος συνάδελφος θα ήθελα να πάρει το λόγο. Uh, Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Κύριος το αναπόφευκτο ερώτημα για το Brexit. Σε ό,τι αφορά του γενικώ τροποποιημένου οργανισμού, υπάρχει ένα σενάριο ότι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί το μονοπάτι των μεταλλαγμένων ε, που δεν ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, εσεί ε, θα μπορούσατε να εικάσετε τι μπορεί να, συμβαίνει, τι μπορεί να σημάνει αυτό Ευχαριστώ κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε μια υποχρέωση από το 2002 για την μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου σε σχέση με τα μεταλλαγμένα. Και υπάρχουν τροπολογίες που έχουν προταθεί. Υπήρχε, κάποια, υπήρξε κάποια τεχνική πρόοδος. Έχουμε την οδηγία το 2010, χωρίς καμιά τροποποίηση. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ, τι προβλήματα υπήρχαν με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερομένους, με τη βιομηχανία. Δεύτερον, μας λέει η Κομισιόν ότι είναι μόνο τεχνικές αυτές οι προσαρμογές, αυτές οι αλλαγές. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούμε στις τελευταίες τεχνολογικέ εξελίξεις. Αλλά εδώ μου φαίνεται ότι υπάρχει και κάτι ακόμη. Η εστίαση υπερβαίνει κατ' την τεχνολογική απλή προσαρμογή. πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της ε, προφύλαξης, αλλά δεν νομίζω ότι καλύπτεται σε όλα αυτά τα στάδια, σε όλες αυτές τις ε, φάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώς έχει μιλήσει και έχει φάσει επιφυλάξεις ε, για τη διαδικασία έγκριση και διοδότηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να δει αυτά τα θέματα Ακούσαμε σήμερα σε μία ακρόαση πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ε, με αυτό το σχέδιο κανονισμού, οδηγίας μάλλον. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι θα καθησυχάσετε πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Χόισλινγκ, ευχαριστώ πολύ. Ούτε κι εγώ ξεκαθαρίσω το μυαλό μου τι λέει η Κομισιόν η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τι θα κάνει, πώς θα μελετά ε, αυτούς τους ε, μεταλλαγμένους ε, οργανισμούς μέσω της νομοθεσίας για τα ζανιοκτώνα ή μέσω αυτής της οδηγίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν είναι τόσο έξυπνο αυτό που προτείνεται κατά την απόψή μου. Νομίζω ότι πρέπει να μας εξηγήσετε πολύ ξεκάθαρα τι ακριβώς προβλέπετε, ποια είναι τα σχέδιά σας. Και ο κύριος Μπαλάς. Ε, ευχαριστώ και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά το νομικό ε, πεδίο που θα επιλέξετε και τι γίνεται σε ό,τι αφορά το προπλασιασμό κλασικών μεταλλαγμένων οργανισμών. Δεύτερο, νέοι γενικώ τοποποιημένοι οργανισμοί. έχουμε αυτά τα νέα υβρίδια και τα λοιπά και θέλουμε να δούμε αν θα ταξινομηθούν ε, μεταξύ των γενετικών στοπημένων οργανισμών ή όχι. Και γίνεται μάχη. Πού βρισκόμαστε ε, σε επίπεδο ΕΦΣΑ όσον ε, αφορά τον επιστημονικό ορισμό των υβριδίων αυτών. Επίσης, υπάρχουν οι ρυθμιστικές απαιτήσει και εδώ στρέφουμε στην Κομισιόν σήμερα. Πού βρισκόμαστε Δεν έχω κάποιον άλλο στον κατάλογο μου, λέει ο πρόεδρος. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν καταρχάς και μετά στον πρόσωπο της ΕΦΣΑ. Παρακαλώ, αν θέλετε, απαντήστε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να απαντήσω. Νομίζω ότι θα πρέπει για μια ακόμη φορά να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που ζητήθηκε ε, από την Κομισιόν. Τι της αναθέσατε να κάνει η Κομισιόν. Όπως είπα εδώ, ανταποκρινόμαστε στην νομική υποχρέωση, δυνάμει το άρθρο 3 της οδηγίας 18 ε, του 2001. Ήταν σαφές, ε, ήταν σαφής εντολή μας, αλλά και πολύ περιορισμένη δυνάμη αυτής της ε, ε, διάταξης για την επικαιροποίηση των παραρτημάτων και την ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών που τότε ίσχυαν στην ΕΦΣΑ. Συγκεκριμένα κατευθυντήρια γραμμή του 2010 που έπρεπε να ενταχθεί όπως επίσης και εξολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων σε σχέση με γενικώ αποποιημένα φυτά. Νομίζω ότι με αυτό απαντώ σε αρκετά από τα ερωτήματα που λένε ότι ίσως η πολύ περιορισμένη στοχευμένη αυτοτροποποίηση από αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία ή ότι δεν λαμβάνει υπόψη νέες ενδεχομένως εξελίξεις ή νέες ε, τεχνικές ε, καλλιέργειας ε, ή χρησιμοποιήσει γενικώς των ποινών οργανισμό. Μην με παρεξηγήσετε όμως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πολύ ξεκάθαρη περιορισμένη εντολή και αυτό έφερε σε πέρας. Υπάρχει και το άρθρο 27 που και αυτό μας περιορίζει. Δηλαδή, εδώ μας ζητείτε μόνο να προσαρμοστούμε στην τεχνική πρόοδο. Κάποια κράτη, μάλλον κάποιοι βουλευτές θα ήθελαν να γίνει μια ευρύτερη τροποποίηση οδηγία ότι θα ήταν κάτι τέτοιο σκόπιμο και επίκαιρο, αλλά δεν ήταν αυτή η εντολή που πήραμε εμείς, δυνάμει αυτή τη διάταξη. από τον Απρίλιο του 2017. Τώρα, να επανέλθω στον χρόνο που χρειάστηκε. Η εντολή μας έλεγε να έχουμε δράσει μέχρι την 3η Απριλίου του 2017. Και αυτό κάναμε. Τότε παρουσιάσαμε την πρόταση και έκτοτε κάνουμε τα διαδικαστικά. Συζητήσαμε και με τα κράτη-μέλη σε μόνιμες διευθυντικές επιτροπές. Αυτό ήταν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ευθύς εξ αρχής. Και εν ώψη της καθοδήγησης ε, του 2010 από πλευρά ΕΦΣΑ, δεν είχαμε άλλες δυνατότητε. Ήταν στενά τα περιθώρια μέσα στα οποία χρειάστηκε να εργαστούμε και για να καταθέσουμε αυτή την τροποποίηση. Έγινε μια παρατήρηση ότι αυτή η τροποποίηση δεν είναι απλή τεχνική τροποποίηση, αλλά κάτι παραπάνω. Εγώ μπορώ να σας πω περισσότερα για τις τεχνικές τροπολογίες. Ε, σας είπα ότι παίρνουμε τα βασικά στοιχεία του εγγράφου της ΕΦΣΑ του 2010, που λέει για μια μεθοδολογία σε έξι βήματα για την αξιολόγηση των κινδύνων των ε, γενετικών στροποποιημένων οργανισμών. Και επίσης ε, έτσι απαντώ στον κύριο Χόισλινγκ που με ρωτάει πού βρίσκεται τελικά η μελέτη αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Πού γίνεται, με βάση τι. Ναι, είναι νομοθεσία για γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς η βάση. Και μέσα σε αυτή την επιστημονική αξιολόγηση του φυτού που υποβάλλεται στην ΕΦΣΑ για εξέταση. Αυτό που έλεγα εγώ, που υπονόησα, είναι ότι αυτή η αξιολόγηση κινδύνου της χρήσης ενός ζανοκτώνου, ενός φυτοφαρμάκου για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, το συγκεκριμένο φυτό, θα γίνει πολύ πιο αναλυτικά από ότι στο πέστος νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα ή τα αυτοπροστατευτικά προϊόντα. όπου λαμβάνονται υπόψη συνθήκε στι οποίε θα καλλιεργηθεί το προϊόν στα μελη το φυτό αυτό στα κράτη-μέλη. Έχουμε και την οδηγία, υπάρχει το opt-out, η πιθανότητα opt-out για τι καλλιέργειε, άρα περιορισμένα τα κράτη-μέλη. Κατά ψευθανότητα που θα επιλέξουν την καλλιέργεια. bulk of the environmental risk assessment as concerns the Όπως είπα, λαμβάνουμε υπόψη μας τις, τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς και επάνω εκεί βασίζεται η αξιολόγηση κινδύνων. Και σε δεύτερη φάση υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει για δεδομένα τα οποία αφορούν τα αυτοπροστατευτικά προϊόντα που σχετίζονται με συγκεκριμένο τροποποιημένο φυτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια καλλιέργεια ανθεκτική στη, στα αυτοφάρμακα που να έχει εγκριθεί και να καλλιεργείται κάποιο τέτοιο φυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Είπε και σε προηγούμενους γραμματείς της ΕΦΣΑ ότι τα μέτρα διαχείριση κινδύνων για τη χρήση του φτωφαρμάκου μπορούν να αποφασιστούν και να αξιολογηθούν στην φάση της άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος, της έγκρισης, της αντιδότησής του. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το πεδίο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το άρθρο 3 της Οδηγίας 18.001 που λέει ποιο είναι το πεδίο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι το πλαίσιο και ποια είναι τα στοιχεία της κατευθυντήριας γραμμής της ΕΦΣΑ. Και επαναλαμβάνω, είναι τεχνική η επικαιροποίηση της νομοθεσίας. Ακριβώς όπως προέβλεπε εντολή μας, δυνάμει του άρθρου που σας προανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σταραθώνα. Thank you very much. I'm a scientist, so I will not be... Πρόεδρε, είμαι επιστήμονας, άρα τα πιο πολιτικά θέματα δεν μπορώ να τα απαντήσω. Μόνο όσα έχουν επιστημονικό περιεχόμενο. Και νομίζω ότι αυτό περιμένει από την ΕΦΣΑ και το Κοινοβούλιο. Για την επιστημονική αξιολόγηση. Επιβεβαιώνω ότι και για τα γενετικά τροπεποιημένα καλλιέργεια σε άλλους οργανισμούς, αλλά και για τα στιζανιοκτώνα. Υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση που ανάγεται στους διάφορους κανονισμούς στην νομοθεσία, ανεξάρτητη αξιολόγηση που είναι αξιολόγηση κινδύνου, που στηρίζεται ειδικά στους όρους χρήσης. Και ε, μιλούμε για τον κίνδυνο από τα ζωνοκτώνα σε γενετικά τροπημένους οργανισμούς, που όμως αναφέρεται όχι στον ε, γενετικά τροπημένο οργανισμό, αλλά στο ζενεοκτόνο το ίδιο. Δηλαδή αυτό θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το ζενεοκτόνο, αλλά και από τις ιδιότητες του ζενεοκτόνου, τις οποίες ιδιότητες για την, επιμερούς, για την ουσία την αξιολογεί η ΕΦΣΑ, ενώ ε, την χρήση την αξιολογεί το κάθε κράτος. Και άρα έχει νόημα να γίνεται η περιβαλλοντική αξιολόγηση της χρήσης του ζυζανιοκτώνου ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβατική καλλιέργεια ή γενετικά τροποποιημένη. Γιατί υπάγεται στον κανονισμό για τα ζυζανιοκτώνα. Δεύτερο στοιχείο. Άλλες εναλλακτικέ για γενετικές τροποποίησεις. Βεβαίως την απόφαση και τον κανονισμό θα του πάρουν το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή του Συμβούλου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή θα αποφασίσουν ε, ποιοι οργανισμοί θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη μεθοδολογία εγκρίνεται ως αποδεκτή. Και εμείς είμαστε έτοιμοι από πλευράς μας για την αξιολόγηση του κινδύνου ή άλλων εναλλακτικών σε περίπτωση που ε, προβληθούν από τους ε, νομοθέτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το θέμα αγαπητοί συνάδελφοι. Και πάμε στο επόμενο. Ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο κατεξουδότησης συμπράξης για τα επιστημονικά κριτήρια τα σχετικά με τους αντοκρινικού διαταράκτες. Ο κύριος Πέραντε εκπροσωπεί την Επιτροπή. Εδώ είναι. Έχετε λόγο για το πολύ 15 λεπτά. Παρακαλώ. Thank you, uh, Madam Chair. Um, uh, the, draft delegated act. Uh... Πρόεδρε, η κατεξότηση πράξη που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά την ε, υλοποίηση υποχρέωση της, της Επιτροπής που απορρέει από το άρθρο 5.3 του κανονισμού για τα βιοκτώνα, πρόταση δηλαδή κριτηρίων για τον εντοπισμό ουσιών με χαρακτήρα ενδοκρινικής διατάραξης, ιδιότητες ενδοκρινικής διατάραξης που θα πρέπει να ε, αντικαταστήσει τα ενδιάμεσα κριτήρια που έχει ήδη προσδιορίσει και προσδιορίζει μέχρι τώρα ο κανονισμός, τα προσωρινά κριτήρια. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη ρήτρα του άρθρου 5, η οποία προσδιορίζει κριτήρια αποκλεισμού όταν ενεργός ουσία δεν μπορεί να εγκρίνεται για χρήση σε βιοκτώνα, μεταξύ των οποίων είναι και αυτές οι οποίες έχουν ε, ιδιότητες ενδοκρινικής διατάραξης για την ανθρώπινη υγεία. Προτείνει λοιπόν την κατεξουσιοδότηση πράξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από διαβουλεύσεις, ευρείες διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων πάντα βέβαια συγκαταλεγόταν και ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επίσης προτιμήσαμε να υποβάλουμε όχι μόνο κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό των ουσιών που μπορεί να έχουν ε, ιδιότητες διατάραξης ενδοκρινικής για τον άνθρωπο, αλλά και αυτών που μπορεί να έχουν ε, χαρακτήρα ιδιότητα διατάραξης ε, του περιβάλλοντος. Αυτό για λόγους αφήνειας. Έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί, οι εταιρείε που εμπλέκονται, που παράγουν, που ζητούν την αδειοδότηση, αλλά και οι αρχέ των κρατών μελών που προβαίνουν σε αυτή την αξιολόγηση και έγκριση, να έχουν πλήρη στοιχεία και τεκμηρίωση στα χέρια του και άρα περισσότερη δυνατότητα πρόβλεψης ε, των εξελίξεων σε σχέση με τα όσα προβλέπει ο τωρινό κανονισμό που δεν δίνει κριτήρια αξιολόγηση συνεπειών στο περιβάλλον. Επίση μπορώ να υπογραμμίσω ότι κατά την πρόταση του κατεξουδότησης αυτού, του κανονισμού, ε, της διάταξης αυτής κατεξουδότησης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα μεριμνά για την περιγραφή κριτηρίων εντοπισμού των ε, ενδοκρινικών διαταρακτών μέσα από τον κανονισμό για τα συζανιοκτώνα, που θα θυμάστε βέβαια και εσείς καλά, τη συζήτηση αλλά και όλη την ψηφοφορία που έλαβε χώρα μόλις πριν από μερικές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Οι προτάσεις είναι ταυτόσιμες ως προς το περιεχόμενο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ενεργές ουσίες είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε βιοκτώνα είτε σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Δεν έχει νόημα δηλαδή να ορίσουμε διαφορετικά κριτήρια για την ίδια ουσία όταν αυτή περιγράφεται ως ενδοκρινικός διαταράκτης ενώ σε άλλη περίπτωση δεν θα, δεν θα καταλήγει τελικά να περιγράφεται ως ενδοκρινικός διαταράκτης. Τα κριτήρια είναι τα ίδια λοιπόν με αυτά του κανονισμού των ζυζανιοκτώνων. Σημαντικό επίσης πιστεύω είναι να υπογραμμίσουμε ότι λόγω του, ε, των διαφορών στο κανονιστικό πλαίσιο, στον κανονισμό για τα βιοκτώνα, η Προποθέσει έγκριση ή μη στοχεύουν ιδιαίτερα στην δημόσια υγεία. Και επιπλέον υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν κατ' εξαίρεση την έγκριση ουσιών που έχουν χαρακτηριστεί, αναγνωριστεί ως ενδοκρινικοί διαταράκτες μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ε, εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον κανονισμό για τα ζυζανιοκτώνα. Κατά τη γνώμη μας, τα κριτήρια συνιστούν σαφή πρόοδο σε σχέση με τα προσωρινά κριτήρια, γιατί τα προσωρινά εκείνα κριτήρια δεν ήταν πρόσφορα. Δεν φέρνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μπορεί να εντοπίσουν δηλαδή και να ταυτίσουν ως ενδοκρινικό διαταράκτη μια ουσία που δεν είναι τελικά πράγματι διαταράκτης, ενώ μπορεί να τους ξεφύγει κάποια άλλη που έχει συνέπειες ενδοκρινικής διατάραξης. Και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτή η κατεξουδότηση πράξη με τα νέα κριτήρια, ε, το ταχύτερο δυνατό, γιατί θα σημάνει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι τα κριτήρια, τα προτινόμενα κριτήρια προστατεύουν τη δημόσια υγεία, προστατεύουν το περιβάλλον, στηρίζονται σε ορισμούς και αρχές σύμφωνους με τις κατευθείαν γραμμές και γενικότερα την περιβαλλοντική νομοθεσία, την νομοθεσία για τη δημόσια υγεία, στηρίζονται σε ευρέως αποδεκτούς ορισμούς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για το τι, ποια, τι σημαίνει ενδοκρινικός διαταράκτης. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντοπίζουν γνωστούς αλλά και ε, ε που για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να έχουν ε, ε, στα συνέπεια δοκρινική διατάραξη στον άνθρωπο αλλά και στο ζώο. Γιατί ό,τι είναι ενδοκρινικός διαταράκτης για το ζώο θεωρείται ότι είναι και για τον άνθρωπο εκτός και να έχει αποδειχθεί ρητά το αντίθετο. Άρα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον κανονισμό των καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών αναπορογωγής ουσιών ακολουθούμε μια προσέγγιση με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, τις επιστημονικές γνώσεις, αντίστοιχα με τα άλλα στοιχεία κινδύνου της, ε, του κανονισμού για τα καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα και τοξικά του, γενε, του αναπαραγωγικού συστήματος. Καταγράφουμε αρνητικές συνέπειες στο ενδοκρινικό σύστημα, σημειώνοντας βεβαίω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει η πειραματική αξιολόγηση της διατάραξη του ενδοκρινικού συστήματος. Δηλαδή έχουμε ευρύτερη ε, προσέγγιση από αυτήν ή αυστηρότερη αν θέλετε προσέγγιση από αυτήν της ε, αιτιολογικής συνάφειας που απαιτεί η Παγκόσμια Οργάνωση απαιτει η παγκοσμια οργανωση Υγεία. Ε, υπάρχει μια αναφορά στο αν χρειάζεται ρητά να αναφερθούμε και σε δεδομένα από άλλες ουσίες. όταν χαρακτηρίζουμε μια συγκεκριμένη ουσία. Έχει και αυτό περιληφθεί στον κανονισμό, τον κατεξουσιοδότηση, διότι οι προϋποθέσεις για τα δεδομένα της, ε, του κανονισμού για τα βιοκτώνα ε, ήδη προβλέπει το σύστημα Reader Cross και άρα ακολουθούμε αυτό το σύστημα. Χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση στάθμισης δεδομένων και άρα μπορούμε να έχουμε χρήση και αξιοποίηση δεδομένων και για, που υπάρχουν ήδη για άλλε ουσίες. Ένα σημείο που πρέπει επίσης να αναφέρω που έχει να κάνει με την προετοιμασία αυτής της ε, διαδικασίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ουσίες είτε ενεργές είτε ε, μέρη ε, μειγμάτων ή άλλων προϊόντων στα οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένε ενεργέ ουσίε. Αυτό ε, είδε κάποια αντίδραση, γιατί κάποιοι, ιδιαίτερα από την παραγωγή, θεωρούν ότι θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ενεργοουσία ενέργεια επιτροπή. Εμεί θεωρούμε ότι ε, η εντολή μα επιτρέπει να συζητούμε και να εξετάζουμε ως διακτάράκτε διακταράκτες ύποπτες ε, όχι μόνο αυτόνομες ουσίε, αλλά και τα μείγματα και θα ήταν παράλογο τα κριτήρια να ισχύουν μόνο για τις ενεργέ ουσίε αλλά όχι για ε, μείγματα ή άλλα προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται αυτές οι ουσίες παρότι θα έχει πάλι τον ίδιο χαρακτήρα διατάραξης το προϊόν. Αυτά έχω να πω ως παρουσίαση. Βεβαίως είμαι στη θέση σας για ερωτήσεις ή σχόλια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για ερωτήσεις. Πείτε μου αν ενδιαφέρεστε αν λάβετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, κύριε είδα. Ναι, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και τις εξηγήσεις. Ήμουν στη μειοψηφία την περσμένη εβδομάδα στην ψηφοφορία και εξέφρασα τη λύπη μου. Ρωτάω τώρα, επειδή θέλω πληροφορίες. Τι γίνεται με τις χώρες μέλη, γιατί ξέρουμε τι δυσκολίες έχουν με τους γάμματα φόμικρον και τις διαφορετικές θέσεις των χωρών μελών. Προτείνει η Κομισιόν, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει από ό,τι φαίνεται, αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά στο θέμα των γάμματα φόμικρον. Ρωτάω λοιπόν την Κομισιόν τι γίνεται με το Συμβούλιο. Έχουν αλλάξει οι θέσεις των μελών μπορούμε μια μέρα να καταλήξουμε σε μια μουσιώδη θέση ενιαία της Ένωσης για αυτούς τους οργανισμούς ή θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Ευχαριστώ κύριε Κουταλάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Κομισιόν. Μια απλή ερώτηση. Αυτή η κατεξουσιοδότηση και ευχαριστω την κομισιον μια απλη ερωτηση αυτη η ερωτηση πραξη πώς επηρεάζει την απαγόρευση πώλησης αυτών των διαταρακτών σύμφωνα με το 19-14 του κανονισμού για τα υποπροϊόντα. Αν λοιπόν η κατοξιοσυδότηση εφαρμοστεί θα συνεχίσει να ισχύει απαγόρευση. Επειδή είχατε μια παρέκκληση η οποία αφορά ενδοκρινικούς διαταράκτες για μη φυσικούς οργανισμούς μια ξεκαθαρή ερώτηση αυτή και θέλουμε ξεκαθαρή απάντηση από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κυρία Κέρλινγκ. Ναι, ευχαριστώ. Τα επόμενα βήματα, να ρωτήσω εγώ. Επαναλημμένως άκουσα από την Κομισιόν ότι θα μπορούσα να δράσουν μετά από την ψηφορία, αλλά μπορούν να το επανεξετάσουν αυτό. Να πω την ανησυχώ για τις προθεσμίες και τις καθυστερήσεις σε σχέση με τον να υπόψη μας τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και για κατά πόσο θα μπορούσαμε ακριβώς να βάλουμε περιθώριο εφαρμογής νέων επιστημονικών δεδομένων. Επειδή και αυτό σε τη θέση μου την ε, προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσαμε να έχουμε λάθος ενδείξεις και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Οπότε αναρωτιέμαι πώς θα αναπτύξει η Κομισιόν κάποια οροζόντια κριτήρια στις διάφορες νομοθεσίες, στους διάφορους νόμους, ώστε να κατανοήσουμε ακριβώς την περιπλοκότητα των νόμων αυτών. Έχετε κάποιο λοιπόν σχέδιο για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Τι να προσδοκάμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Κομισιόν επίσης. Όπως ξέρετε είχα μια ανυποχώρητη θέση για αυτά τα θέματα. Απορρίψαμε την απόπειρα της Κομισιόν να θεσπίσει παρεκκλήσεις οι οποίες δεν επίπτουν στο πεδίο του κανονισμού και μία ερώτηση σχετικά προς την Κομισιόν. Τι θα κάνει η Κομισιόν για τα βιοκτώνα και τη στιγμή μάλιστα που θα έχουμε σοβαρές αποκλήσεις μεταξύ κανόνων και κριτηρίων για βιοκτώνα και ζανιοκτώνα. Και το Κοινοβούλιο επίσης επανειλημμένως έκανε έκκληση για σωστά οριζόντια επιστημονικά κριτήρια και το τι αποτελεί ενδοκρινικό διαταράκτη σε σχέση με την προστασία της μόσιας υγεία και του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε πάντως να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με το σχέδιο κατοξιδότησης πράξη ε, πράξης για τα βιοκτώνα σε σχέση με, τα, με τις αποδείξεις, το βάρος των αποδείξεων. Δηλαδή, τι γίνεται με τις παρενέργειες αυτών των διαρακτών, διαταρακτών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει η Κομισιόν πώς θα προχωρήσει, ποια προσέγγιση θα ακολουθήσει και πώς θα δικαιολογήσει αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζενκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε τα κριτήρια για τα ζυζανιοκτώνα στο Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπαναχωρήσει και θα υποχωρήσει μάλλον στις πιέσεις των λόμπι και θα επιτρέψει να επανέλθουν το παράθυρο από την Κομισιόν αυτά τα κριτήρια. Το ίδιο και για τα βιοκτώνα. Αυτά που γίνονται εδώ να ακατανόητα για μένα και θεωρώ ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ακούσει αυτούς που σύμουν τον κόδωνα του κινδύνου για τους διαταράκτες. Εσείς υποβάλλετε μια πρόταση όπου παρεσφρίουν από το παράθυρο πάρα πολλέ ουσίες και μου φαίνεται παράδεκτο αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Γκροστέτ είπε προηγουμένως, η κυρία Τελάκ, ότι εμείς δεν συμφωνήσαμε με τις αντιρρήσει. Γιατί καλύτερο να έχουμε μια τελή νομοθεσία από το να μην έχουμε καθόλου. Ιδιαίτερα όσον αφορά την τονή κατάσταση αυτών των διαταρακτών. Εγώ λοιπόν ανησυχώ σε σχέση με την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας, επειδή τίποτα δεν τους προστατεύει σήμερα από αυτούς τους αντοκρινικούς διαταράκτες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει η Κομισιόν ποιες είναι οι άμεσες προοπτικές, όχι σε λίγα χρόνια, άμεσα, αύριο, τι μπορούν να κάνουν ώστε να προστατεύσουμε τους συμπολίτε μας και την υγεία τους. Εδώ κλείνει ο κατάλληλος των ομιλητών που είχα. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι. Αν όχι, στρέφομαι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πέριν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τους βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Να ξεκινήσω με το ερώτημα της κυρίας Γκροστέτ για την ε, κατάσταση στα κράτη-μέλη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το, το Συμβούλιο φαίνεται ότι θα αποφασίσει να μην προβάλλει ένσταση σε αυτή την κατεξοδότηση πράξη για τα κριτήρια στο πλαίσιο των, του κανονισμού για τα βιοκτώνα. Αυτό σημαίνει ότι από πλευρά Συμβουλίου δεν υπάρχει αντίρρηση για την έναρξη ε, ισχύω αυτή τη κατεξοδότηση πράξη όπω την ε, κατέθεση Κομισιόν. Το ερώτημα που έχει να κάνει με τον αντίκτυπο των προτινόμενων κριτηρίων στο άρθρο 19.4 Δέλτα που λέει ότι απαγορεύεται η πώληση βιοκτώνων που έχουν ιδιότητες ανδοκρινικού διαταράξη στο, γενι... στο πλατή κοινό. Να απαντήσω, επειδή ήταν πολύ άμεσο το ερώτημα, με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι ακριβώς η ρήτρα που ε, κίνησε και την αντίρρηση προηγούμενη εβδομάδα ισχύει ε, και στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή για την ε, αναγνώριση των ενδοκρινικών διατακτών σε σχέση με τη δράση του προ το περιβάλλον και ιδίω μειωμένων αριθμό μικροοργανισμών μη στόχου. Στη παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα το είπα και μπορώ να το επαναλάβω. Οι ουσίες που καλύπτονται είναι ουσίες που έχουν ένα συγκεκριμένο δρό, τρόπο δράσης ε, μέσω του ενδοκρινικού συστήματος, τα έντομα και η τοξικότητά τους θεωρείται σχετικά θετική. Το άρθρο 19.4 Δέλτα στο BPA δεν αναφέρεται σε ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη για οργανισμούς στόχους ή μη στόχους. αλλά και οι ουσίες που έχουν αυτή τη δράση την ενδοκρινική διατάραξη στα οργανισμούς στόχους, καλύπτει τον τόπο και δραστικές ουσίες που έχουν δράση σε μη στόχους. Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι στις διατάξεις. Το άρθρο 19.4 Δέλτα ισχύει, εφαρμόζεται και τα προϊόντα που έχουν αυτές τις ε, ιδιότητε δεν μπορούν να πολλούνται στο λατικινό. Για την κυρία Γκέρλινγκ και την κυρία Ντελαέ που ρώτησαν ποιε είναι οι προθέσει μα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Θα εξαρτηθεί κατά κάποιο βαθμό από το τι θα συμβεί τώρα εδώ στο Κοινοβούλιο. Τι θα αποφασίσετε για αυτό το σχέδιο κατεξουσιοδότηση πράξη. Και καταρχάς θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μοίρα αυτή τη ε, πράξη και μετά εμεί θα προβούμε σε ε, προβληματισμό κατά πόσο θα καταθέσουμε άλλες προτάσεις ε, για τα κριτήρια κλινικών τεταρακτών στο πλαίσιο των ζυζανιοκτώνων. Συμφωνούμε με την επιθυμία που εξάφησαν ορισμένοι ομιλητέ ότι θα πρέπει να είναι συνεκτικά κριτήρια τα οποία θα ισχύουν για όλου το ίδιο και το πώ θα προχωρήσουμε θα εξαρτηθεί, όπω είπα, από το τι θα συμβεί σε αυτή την καθεξουσιαδότηση πράξη ευρύτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ήδη ότι θα προχωρήσει σε μια πρόταση για μια νέα στρατηγική στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Είναι όμως ακόμη πρόωρο το στάδιο, είμαστε στη φάση του προβληματισμού. Θα δούμε τι θα γίνουν αυτά τα κριτήρια και τα κριτήρια για, το, για τα ζανιοκτώνα, γιατί αυτό θα επηρεάσει και τον προβληματισμό μας εν γέννη. Φυσικά και εμείς συμφωνούμε με την επιθυμία που εξέφασε η κυρία Γκέρλινγκ, σε ό,τι αφορά τα ενδιάμεσα, τα προσωρινά κριτήρια για βιοκτώνα και ζυζανιοκτώνα, να αντικατασταθούν τα κατάλληλα κριτήρια με κριτήρια που θα είναι κατάλληλα και τα ενδεδειγμένα για την προκειμένη περίσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη κυρία Νταλή Χάζεκαμπ, που λένε ότι η πρότασή μα κατά την άποψή του δεν είναι ενδεδειγμένη, γιατί απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία υψηλού επίπεδου. Εμείς, το είπα και στην εισαγωγή μου, διαφωνούμε. Το επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων που απαιτείται είναι απόλυτα συγκρίσιμο με αυτό που απαιτείται για άλλε ε, σημαντικέ ε, καταστάσεις ε, επικίνδυνες όπως είναι οι μεταλλαξιογόνες, τοξικές κτλ. ιδιότητες. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να ισχύει συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Άρα αυτή η αξίωση, αυτός ο ισχυρισμό ότι τα κριτήρια προτείνονται, απαιτούν πολύ ε, σημαντικά ε, αποδεικτικά στοιχεία, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Προτείνουμε την υποβολή αναφορών και αξιολόγηση ε, που υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνεται μετά από 7 χρόνια το πολύ. Μπορεί να γίνει και νωρίτερο όμως αν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια. Δεν το πιστεύουμε βέβαια εμεί. γιατί πιστεύουμε ότι ό,τι έχουμε προτείνει ευθυγραμμίζεται απολύτω με τα απαιτούμενα για άλλε επικίνδυνε ουσίε και μα επιτρέπει νομίζω να πετύχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασία τόσο τη ανθρώπινη όσο και του περιβάλλοντο. Ευχαριστώ. Είναι νωρί, λέει πρόεδρο. Έχω να δώσω τώρα στην κυρία Κούτελα που θέλει να κάνει μία ακόμη ερώτηση. Ναι, για εσά είναι η ερώτηση ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις πολύ σαφείς απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις για αυτή την απαγόρευση που ισχύει από ό,τι φαίνεται και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι. Εσείς ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος να φροντίσετε να έχετε γραπτός τη σαφή απάντηση που πήραμε προφορικά σήμερα από την Κομισιόν. Να ζητήσετε γραπτός αυτή την επιβεβαίωση. Αυτό είναι το αίτημά προς εσάς κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η ευχαριστώ πολύ κύριε Κούτελα, το σημείωσα. Ε, θέλω να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ε, ολοκληρώσαμε νωρίς νωρίς, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τι ώρα στις 9, 9 το πρωί. Γεια σας.